Σας ζητώ εκ νέου συγγνώμη που χρειάστηκε να απουσιάσω. Ξαναρχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Βεβαίως, καταρχάς, με τις ανακοινώσεις του Προέδρου μετά την συνεδρίαση των συντονιστών. Για την τροποποίηση του κανονισμού εγώ θα είμαι ο εισηγητής ε, και θα σας μιλήσω για τις, τα συμπεράσματα. Επίσης, αν συμφωνείτε, θα ήθελα να ζητήσουμε την νομική γνωμοδότηση για το θέμα της εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 48 του, της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας σε περίπτωση που αποχωρήσει η Σκοτία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει ένα έγγραφο που στείλαμε στην ε, κυβέρνηση της Σκοτίας και αποφασίσαμε για αυτό το θέμα να ζητήσουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Προτείνω δηλαδή να εγκρίνεται αυτό το αίτημα. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στη Ρώμη 24 με 26 του μηνός από μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας, οι συντονιστές σημείωσαν ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να έχει η αποστολή αυτής της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 7 μέλη και προτείνουν δύο από το ΕΛΚ, ένα από τους σοσιαλιστές, ένα από το, τους πράσινους, ένα από το ECR και ένα από τους φιλελεύθερους. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και βλέπω ότι δεν υπάρχουν, νομίζω ότι εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Πάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 136 του κανονισμού για τη συμμετοχή των ε, βουλευτών στις Ολομέλειες. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ που είναι ο εισηγητής. Έκανα λάθος το όνομα, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Χέφνερ, συγγνώμη. Ο κύριος Χέφνερ ζήτησε να κάνει μια σύντομη παρέμβαση πριν την ψηφοφορία. Παρακαλώ κύριε Χέφνερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρωτού αρχίσει η ψηφοφορία, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία άσκηση, μία άσκηση για την διαδικασία και τον κανονισμό, τον εσωτερικό κανονισμό. Ο εσωτερικός κανονισμός αυτή τη στιγμή προβλέπει τα μέλη του Κοινοβουλίου να δικαιολογούνται όταν απέχουν από κάποια συνεδρίαση, για παράδειγμα για άδεια μητρότητας, όταν υπάρχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, ασθένεια ή ε, σημαντικές αποστολές. Όμως, στο πρωτόκολλο καταγράφονται ως απόντες, αδικαιολόγητοι. Και αυτό χαροποιεί πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης όταν ε, αναφέρονται στους ε, ευρωβουλευτές, στις απουσίες, στο ότι λείπουν από τις συνεδριάσεις των επιτροπών. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι όταν ε, πραγματικά υπάρχει σοβαρός ο λόγος για να λείψει κάποιος ευρωβουλευτής να ε, σημειώνεται αυτό στα πρακτικά. Ε, σε αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι και επίσης έχουμε συμφωνήσει σχετικά με τις άδειες μητρότητα στον εσωτερικό κανονισμό να αναγράφονται και οι άδειες πατρότητας. οι γονικές άδειες δηλαδή. Αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον εσωτερικό κανονισμό και θέλουμε να... Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 31 του εσωτερικού κανονισμού, θέλουμε όμως να διευκρινιστεί το σημείο αυτό. Εξού και η παρέμβασή μου λοιπόν. Αφότου ψηφιστεί η έκθεσή μου, θα μπορούσε ο πρόεδρος της Επιτροπής να στείλει μια επιστολή στο Προεδρείο με την παράκληση να διευκρινιστεί στα εκτελεστικά μέτρα του άρθρου 31 τι είναι η άδεια μητρότητας, πατρότητας, γονική άδεια και να ληφθούν αυτά υπόψη για τις παρουσίες των βουλευτών και καθώς επίσης και η υιοθέτηση ενός παιδιού και η άδεια, η γονική άδεια μετά την υιοθέτηση ενός παιδιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στη ψηφοφορία λοιπόν. Έχουμε μία τροπολογία, την ε, τροπολογία 1 του εισηγητή. Παρακαλώ, όποιος είναι υπέρ να σηκώσει το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αποχές. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση. Ποιος είναι υπέρ, να σηκώσει το χέρι παρακαλώ, της έκθεσης. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον κύριο Χέφνερ. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση Γκουρμάη για την τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού σχετικά με τις κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις. Θα ήθελα η Αντιπρόεδρος Γκουρμάη να αναλάβει την Προεδρία για μία στιγμή, γιατί πρέπει να απουσιάσω. Αν μου επιτρέπετε θα απουσιάσω για λίγο. Ευχαριστώ. Είχα καθυστέρηση γιατί ήμουν στην Επιτροπή Μεταφορών. Για την έκθεσή μου, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι λάβατε τις τροποποίησεις που μοιράστηκαν πριν 10 μέρες περίπου. Εγώ υπέβαλα δύο επιπλέον τροπολογίες την περασμένη εβδομάδα, λίγο αργότερα δηλαδή. Όλες οι τροπολογίες ευθυγραμμίζονται μετά όσα συζητήσαμε το Δεκέμβριο στην Επιτροπή, στην προηγούμενη ανταλλαγή των απόψεων. Ήταν πολύ καλή αυτή η συζήτηση, ζωτική σημασία. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας τότε. Έχω 18 νέες τροπολογίες συνολικά στην αρχική μου έκθεση που καλύπτει το θέμα του άρθρου 180 για τις γραπτέ γραπτές ερωτήσεις. Τώρα για το χρόνο μιλίας. 117. Το θέμα είναι τι γίνεται με την κάλπη, ότι πρέπει να βρίσκεται εκτός του χώρου της Ολομέλειας ούτω ώστε να μην διαταράσει την διαδικασία των συζητήσεων. Για τις ε, γραπτές ερωτήσει, συγγνώμη, 118 είναι το άρθρο αυτό, σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές με την ε, Κομισιόν και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, το θέμα είναι να μην υπάρχουν καταχρήσεις και έχω προβλέψει τους τρόπους με του οποίου θα αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση, γιατί οι βουλευτέ με τι γραπτέ ερωτήσει απλώ ασκούν τον έλεγχο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τι γραπτέ ερωτήσει για να κάνουμε πολιτικέ δηλώσει. Δεν θα πρέπει να τι χρησιμοποιούμε για να δημιουργούμε, για να φτιάχνουμε στατιστικέ, οι οποίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λάθο τρόπο ε, για να αξιολογηθεί ο τρόπο με τον οποίο δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό το στόχο, οι τροπολογίε που υπέβαλα ε, στηρίζω, ε, εστιάζουν σε τρει τομείς, ε, σε τρεις περιοχές. Ε, να εξουσιοδοτήσουμε το Κοινοβούλιο, τον Πρόεδρο και την υπηρεσία του να παίρνει αποφάσεις για την, ε, το παραδεκτό ή όχι μιας ερώτησης, δηλώνοντας ότι η οχι βασίζεται στον εσωτερικό καονισμό γενικά. Φυσικά, λαμβάνοντα υπόψη το πνεύμα των άρθρων του δηλωνοντας οτι η αποφαση του Προέδρου θα πρέπει να βασίζεται στους, στον εσωτερικό κανονισμό γενικά. Φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα των άρθρων του κανονισμού. Και όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η συνθήκη. Τροπολογία 4, 13 και 20. Μιλάνε για αυτό το θέμα. Επίσης, κάποια όρια θα ήθελα να αναφέρω. Τροπολογία 5. Ε, περιορίζονται οι ηλεκτρονικές ερωτήσεις, 5 το μήνα. Μετά, πάνω από το 5, θα πρέπει η υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αρμόδια να τις αξιολογήσει. Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις α, θα δοκιμαστούν για, μία, για ένα χρόνο και μετά η διάσκεψη των Προέδρων θα αξιολογήσει κατά πόσο πρέπει να συνεχιστεί αυτό το σύστημα. Όπως είπαμε το Δεκέμβριο, αυτή η φόρμουλα ε, έδωσε καλά αποτελέσματα στο House of Commons, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Επίσης, η τροπολογία 19 που υπέβαλα περιορίζει τις ερωτήσεις σε 200 ε, λέξεις, ούτως ώστε να μην γίνονται πολιτικές δηλώσεις, να είναι μια πραγματική δηλαδή η ερώτηση. Και ακόμα μια τροπολογία, η τροπολογία 15, Μιλάει για όριο. Κάθε ερώτηση πρέπει να έχει το πολύ τρει υποερωτήσει. Οι στατιστικέ ερωτήσει θα πρέπει να πηγαίνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι η υπηρεσία έρευνα. και να αποφύγουμε τι επαναλήψεις παρόμοιων ερωτήσεων, γιατί πιστεύω ότι είχαμε και αυτό το πρόβλημα πολύ συχνά. Πιστεύω ότι αυτέ οι διαφορετικέ τροπολογίε θα βοηθήσουν σημαντικά να μειώσουμε τον αριθμό των περιττών ερωτήσεων ούτω ώστε οι βουλευτέ να μπορούν να χρησιμοποιούν 100% το δικαίωμά του να, ασκούν πραγματικές, να υποβάλουν πραγματικέ ερωτήσει. Είμαι φυσικά ανοιχτή για ερωτήσεις στην πρότασή μου. Εάν θέλετε, σηκώστε το χέρι σα, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Ο κ. Ντάβεβε είναι ο πρώτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και η συγγήτρια παράλληλα. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσίαση. Και εγώ έχω υποβάλει φυσικά διάφορες τροπολογίες και είναι παρόμοιες με αυτές που ακούσαμε από εσά, τις δικές σας δηλαδή. Υπάρχει πραγματικά μεγάλη δυνατότητα για συμβιβασμούς. ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα και μια συνένεση. Η τροπολογία 15. Για την τροπολογία 15 να σας πω το εξή. Εξήγησα ποιο, κατά τη γνώμη μου, είναι το σημερινό πρόβλημα στην τροπολογία 15 σε σχέση με τις γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. 32% από αυτές υποβάλλονται από 10 μόνο ευρωβουλευτές, το 32% των ερωτήσεων. Και 45% των ερωτήσεων υποβάλλονται μόνο από 20 άτομα, 20 ευρωβουλευτές. Μάλιστα ένας ευρωβουλευτής υπέβαλε σχεδόν 900 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ορισμένοι ευρωβουλευτές αντί να χρησιμοποιούν το ίντερνετ ή το τηλέφωνο για να βρουν τις απαντήσεις σε απλά ερωτήματα που είναι απλώς πληροφοριακής φύσεως ή τεχνικής φύσεως. Απλώς υποβάλλουν σωρία κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Και πέφτουν βροχή αυτές οι ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Αυτό όμως έχει κόστος αν υποβάλουμε τόσες πολλές ερωτήσεις, πρέπει να κάποιος να τις διατρέξει, πρέπει να απαντήσει. Δεν ξέρουμε το κόστος για την Κομισιόν, αλλά για το Κοινοβούλιο είναι περίπου 4.000 ευρώ ανά κοινοβουλευτική ερώτηση. Η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει σε μία ερώτηση μόνο αν έχει περάσει από τη διαδικασία τη συλλογική του σώματος των επιτρόπων. Και το κόστος για την Κομισιόν είναι σημαντικό. Φυσικά η δημοκρατία έχει ένα τίμημα. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να φημώσουμε αυτούς που πραγματικά επιθυμούν πολιτικές απαντήσεις σε πολιτικές ερωτήσεις αλλά έχω πραγματικά την αίσθηση θα πρέπει να υποβάλλονται ερωτήσεις που έχουν περάσει από αυστηρότερο, αυστηρότερο ποιοτικό έλεγχο. Και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ένα το όριο στον αριθμό των ερωτήσεων που μπορεί να υποβάλει ένας μόνο ευρωβουλευτής. Στο συμβασμό πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε τελικά επακριβώς στον αριθμό των ερωτήσεων που μπορεί να υποβάλει ένα μόνο άτομο. Επίσης, θέλω η διαδικασία κοινοβουλευτικών ερωτήσεων να επεκταθεί και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι ένα παλιό πρόβλημα που είχα Θέλω ο κ. να μπορεί να απαντά κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την προσωπική του ατζέντα. Δεν είναι όμως έτοιμος να απαντήσει σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και, αυτός, και αυτό είναι ένα πρόβλημα και μια έλλειψη. Και θα πρέπει να πιέσουμε τον διάδοχό του που θα διοριστεί ή θα εκλεγεί το φθινόπωρο για να δεχτεί κάτι τέτοιο. Να σταματήσει αυτή η πρακτική και να βελτιωθούν τα πράγματα. Περιμένω λοιπόν τη συνέχεια αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ. Όπως μου είπαν δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά βεβαίως θα δώσω τώρα με μεγάλη χαρά το λόγο στην κυρία Γιαννάκου. Και εν συνεχεία θα ήθελα να κλείσουμε όμως γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Μαριέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας συγχαίρω για την έκθεσή σας Ζήτα. Ε, συμφωνώ με τον Άντριου και με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει ότι ορισμένοι εκμεταλλεύονται και το χρόνο των προφορικών τροπολογιών, ε, ερωτήσεων και το χρόνο των γραπτών. Διότι στα κράτη-μέλη υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες και έντυπα που ασχολούνται με τον αριθμό των ερωτήσεων. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται ορισμένοι να έχουν κάνει απίθανους αριθμούς ερωτήσεων και να εμφανίζονται ως οι καλύτεροι βουλευτές στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, επειδή γίνονται συνεχώς οι ίδιες ερωτήσεις, βέβαια έκθεσή σας αφορά κυρίως τις προφορικές ερωτήσεις, αλλά επειδή γίνονται συνήθως οι ίδιες ερωτήσεις, έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην απαντά επί της ουσίας πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας τρόπος σοβαρής διαλογής για να έχουμε σοβαρό πολιτικό διάλογο. διαφορετικά οι ερωτήσεις έχουν γίνει ένα σύστημα διαχειριστικό τελείως ε, όπου ορισμένοι το εκμεταλλεύονται όπως εκμεταλλεύονται την μπλε κάρτα μέσα στην ολομέλεια κτλ. για να στέλνουν ανακοινώσεις στη χώρα τους. αλλά η δουλειά των ευρωβουλευτών δεν είναι αυτή φυσικά και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι γελιοποιούμεθα θυμάμαι και σε παλιότερες εποχές επί 800 ερωτήσεων τις 500 τις είχαν κάνει δύο άτομα. Κύριε Πρόεδρε πρέπει αυτό να το, να το περιορίσουμε. Δεν μπορεί να γελιοποιούμε. Θα, γελιοποιούμε θα όλοι μαζί με αυτά που γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Θα λάβω υπόψη και τα δύο σχόλια και φυσικά επιθυμώ να οδηγηθούμε όλοι σε κάποια συμβαστική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Γιαννάκου να λάβει ξανά το λόγο. Θα μας ενημερώσει σχετικά με τον τριμερή διάλογο για την έκθεση σχετικά με τα πολιτικά κόμματα. Να σας υπενθυμίσω ότι η... ο ότι στην ε, προηγούμενη συνεδρίαση μάλλον Συναντηθήκαμε και με τον υπεύθυνο Υπουργό για το θέμα αυτό. Κύριε Γιαννάκου, έχετε το λόγο. Λοιπόν, και φυσικά πιστεύω πως ε, θα ήταν πολύ χρήσιμο να είχαμε μια συνάντηση των σχεδόν εισηγητών αύριο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, θα γίνει μια συνάντηση των εισηγητών διότι έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία έρχεται από, το, ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο και επομένως ε, είχα ήδη ειδοποιήσει τη Γραμματεία να συναντηθούμε αύριο, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε, να δούμε το κείμενο αυτό και βέβαια η ελληνική προεδρία θέλω να σας πω ότι επιδιώκει μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου να έχει πάρει full mandate για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στα σοβαρά το σύνολο της ε, πρότασης αυτής το οποίο όπως σας έχω πει πολλές φορές αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον και στα κράτη-μέλη και από τον τύπο. Επομένως θα προχωρήσουμε. Ε, νομίζω ότι έχετε ήδη όλη η, shadows, όλη η διαπραγματευτική ομάδα το κείμενο αυτό το οποίο μας εστάλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα το δούμε αύριο θα γίνει και τεχνικός διάλογος αν χρειαστεί και πάντως ε, έτσι θα προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι θα εξασφαλιστεί τελικά το full mandate από την ελληνική προεδρία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συνεργασία μας και τον τριλόγο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Αντριου Νταφ θα ήθελε να το σχολιάσει. Κάποιος άλλος, κύριε Μπρόντς, σας καταγράφω στο κατάλογο. Νομίζω ήμουν σαφής. Ζήτησα από όποιον θέλει να λάβει το λόγο και δεν το κάνατε. Τέλος πάντων, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Κύριε Ντάφ, αρχίζετε πρώτος. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να πω μόνο ότι ελπίζω η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου να είναι πιο αποτελεσματική στον τριμερή διάλογο από ότι ο προκατοχός της και είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Θα πρέπει να γραφεί στα πρακτικά ότι η προηγούμενη συνεδρίαση του άτυπου τριμερούς διαλόγου το Δεκέμβριο οδήγησε σε μία συμφωνία, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το θεσμικό μέρος του πακέτου. Έχουμε πάρα πολλά σημαντικά, ουσιαστικά θέματα, όμως τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν η πρόοδος που θα γίνει πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρόντς. Ε, ήθελα να πω κάτι για τη δική σας έκθεση. Κυρία Πρόεδρε, αντί να τεθεί ένα όριο, αριθμητικό όριο για τον αριθμό των ερωτήσεων, θα προτιμούσα δημοσιότητα. Δημοσιότητα για εκείνους που περνάνε όλη τους ε, τη ζωή υποβάλλοντας ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν υποβάλει 890 ερωτήσεις. Θα... Με ενδιαφέρε προσωπικά να μάθω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει τόσο μοναξιά, που δεν έχει φίλους και νιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταυτού. Έχετε δίκιο. Πραγματικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να σας πούμε ποιος είναι. Είναι όμως ε, κάτι που κάνουμε ε, σε συνεργασία. Λυπάμαι, λοιπόν, για το επιτελείο του συναδέλφου ο οποίος έχει υποβάλει τόσες ερωτήσεις. Όπως και να έχει όμως, όσον αφορά το δικό μου σχόλιο για τη χρηματοδότηση των ε, πολιτικών κομμάτων, να πω ότι φυσικά ξέρουμε ότι οι προθεσμίες είναι στενές, μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας υπάρχει όμως η δυνατότητα να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και θα πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν τη δουλειά μας και τις προσπάθειές μας. Θα ήθελα να επιμείνω επίσης στο ότι υπάρχει ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο στην ώρα του για τις ε, διαπραγματεύσεις και ο χρόνος κύλα και πιστεύω πως θα χρειαστούμε πολύ περισσότερες ενέργειες πολύ περισσότερη συζήτηση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε το θέμα στα σοβαρά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της Επιτροπής μας αυτής και πρέπει να είμαστε σε θέση να ε, εργαστούμε σε αυτό με μεγάλη ταχύτητα. Ο κύριος ε, Σέφερ τώρα θα ήθελε να κάνει κάποια σχόλια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Και να σας πω και τι είπε η Ελληνική Προεδρία την περασμένη εβδομάδα. Όντως ελπίζουν να έχουν μια πλήρη διαπραγματευτική εντολή, full mandate, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Είναι βέβαια αργά, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει αρκετή αντίσταση από το Συμβούλιο για όλο αυτό το θέμα. Δεν θα είναι λοιπόν εύκολο το έργο μας και πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Σίγουρα όλοι έχουμε εργαστεί σκληρά, αλλά θα υπάρχει μάλλον τόσο μεγάλη αντίσταση από το Συμβούλιο που θα πρέπει να αναβάλουμε το θέμα μέχρι μετά τις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά. Και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρατε αυτό, διότι το κοινοβούλιο είναι τελείως διαφορετικό, μπορεί να μην έχουμε πλειοψηφία. Δεν βλέπω κάποιον άλλο συνάδελφο να ζητά το λόγο. Θα ζητήσω λοιπόν από την εισηγήτρια να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι έχουμε μείνει όλοι σύμφωνοι πρώτον σε αυτά που συμφωνήσαμε το Δεκέμβριο. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση περί αυτού. Υπήρξε ίσως κάποια παρεξήγηση γιατί σε ένα σημείωμα της γραμματείας αναφερόταν απλώς τι είχε πει ο καθένας μας. Αλλά η συμφωνία, κύριε Ντάφ, παραμένει συμφωνία, δεν υπάρχει ε, λόγος ανησυχίας ε, αύριο θα συναντηθούμε θα επικοινωνήσει ε, η γραμματεία για να δούμε ποια είναι η πιο κατάλληλη ώρα για να μπορέσουμε να εργαστούμε μαζί πάνω στο κείμενο που έχει στείλει για το funding για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια και το σύνολο για να είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα, το θέμα που έθεσε ο κύριος Σέφλιν, γιατί όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε, είναι πιθανό να υπάρξει, να συνεχίσει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση μέσα στο Συμβούλιο. Ε, τότε κύριοι συνάδελφοι εμείς οφείλουμε πριν λήξει η θητεία αυτή να το ψηφίσουμε στο κοινοβούλιο. Πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια. Και από εκεί και πέρα τι θα κάνει ε, το νέο κοινοβούλιο αυτό είναι μια άλλη ιστορία δεν ξέρουμε καν πως θα είναι το νέο κοινοβούλιο αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο δεσμευτικό να έχει πάρει θέση συνολικά το κοινοβούλιο και να το ψηφίσει αν η προεδρία δεν καταφέρει αυτή τη συμφωνία μεταξύ μας στον Τρίλογο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι υποστηρίζουμε αυτά που μόλις είπατε συνοψίζοντας. Όταν έρθει ο κύριος Κασίνη, ή μάλλον ο κύριο Κασίνη δεν είναι εδώ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σταματήσουμε για 10 λεπτά. Α, μόλι έφτασε όμω ο πρόεδρο. Μόλι έφτασε. Επομένω, επειδή η έκθεση είναι του κυρίου Κασίνη, να του δώσουμε απλώ ένα λεπτό για να έρθει στην έδρα. Κύριε Κασίνη, η έκθεσή σα. Θα περιμένω να αποφασίσει ο κύριο Κασίνη. As I told you, Mr. Scholz is going to be back uh, only a bit uh, later. Ο κ. Σόλτ δεν θα έρθει ακόμα πιο αργά. Θέλω να πω επίσης ότι ελπίζω πως η γραμματεία μας θα οργανώσει την ε, συνάντηση των σκιωδών για τα πολιτικά κόμματα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση, να φτάσουμε σε μια ενιαία προσέγγιση για αυτή τη θαυμάσια έκθεση. Για να δούμε λοιπόν τι θα αποφασιστεί. Περιμένω λοιπόν να δω και τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος τώρα. Okay, so the final instruction uh, from... Τι είπε ο πρόεδρος. Θα κάνουμε διάλειμμα μισής ώρας. Ζητώ συγγνώμη. Θα σταματήσουμε για μισή ώρα. Άνθρωποι είμαστε. Χρειάζεται μερικές φορές να κάνουμε διάλειμμα. Σε 30 λεπτά ακριβώς θα ξαναρχίσουμε. Ευχαριστώ.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

ποτέ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

Μετά από αυτό το διάλειμμα, ας ξαναρχίσουμε, παρακαλώ, τη συνεδρίασή μας. Εγώ κανονικά μίλαγα προτελευταίως. Η... Το διάλειμμα δεν οφειλόταν στη δική μου απουσία, αλλά ουσιαστικά στην απουσία ενός άλλου συναδέλφου. Επομένως, χρειάστηκε να... χρειάζεται τώρα να αλλάξουμε την ε, σειρά της ε, των θεμάτων της μέσια διάταξης. Πρώτα θα κάνουμε το δικό μου θέμα και μετά το θέμα της Τρόικας. Το δικό μου θέμα είναι οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και για αυτό το θέμα δεν έχω έτοιμη ακόμα την έκθεση, το κείμενο δηλαδή. Θα πρέπει να δουλέψω επίσης πολύ γρήγορα. Η σημερινή μας συνάντηση τι εξυπηρετεί να συγκεντρώσω τις δικές σας παρατηρήσεις. Σήμερα βεβαίως εγώ μπορώ να κάνω μόνο προκαταρτικές παρατηρήσεις. Έχω ήδη εξετάσει πάρα πολλά, πάρα πολλά κείμενα. Έχω κοιτάξει τις παλιές εκθέσεις από τον κύριο Μπροκ, αλλά και από τον σημερινό πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, του, τον κύριο Ναπολιτάνο. Ο Ναπολιτάνο ετοίμασε την εκθεσή το 2002 και ο Μπροκ ε, το 2009. Και υπάρχει μια άλλη έκθεση του 2007. Στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας ε, δημιουργήθηκε μια ομάδα προβληματισμού για να ασχοληθεί με το θέμα των σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δούλεψε για δύο χρόνια και ετοίμασε ένα κείμενο. Όλα αυτά τα κείμενα λοιπόν υπάρχουν, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε ετοιμάζοντα τη, τη δική μου έκθεση. Ειδικά για την έκθεση Ναπολιτάνου, να σα υπενθυμίσω ότι τα βασικά σημεία ήταν όχι στην ιδέα ενό δεύτερου σώματο που θα αποτελείται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, ήταν μια ιδέα μετά το Μάστριχτ, ειδικά στην... Ε, οι Γάλλοι το είχαν προτείνει να δημιουργηθεί ένα δεύτερο πούμε, κοινοβουλευτικό σώμα. Η έκθεση Ναπολιτάνου έλεγε ότι κάτι τέτοιο θα είχε περιπλέξει και θα είχε καθυστερήσει την ε, κοινοβουλευτική διαδικασία. Επίσης έλεγε όχι αυτή η έκθεση στην παρουσία των εκπροσώπων των ε, κοινοβουλίων στο Συμβούλιο μαζί με τους Υπουργούς για να ενισχυθεί ας πούμε η... το δεύτερο αυτό σώμα του Συμβουλίου. Επίσης η έκθεση Μπροκ μιλούσε πολύ για τη σημασία του πολιτικού ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια των κυβερνήσεών τους με τρόπο πιο αποτελεσματικό, ούτω ώστε να συμμετάσχουν στην ε, οικοδόμηση της Ευρώπης. Και τονίζει ότι θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να συνεργαστούν για την μεταφορά των ευρωπαϊκών κανόνων σε εθνικό επίπεδο και την ασωμάτωσή του στην εθνική νομοθεσία. Όλα αυτά τα διαβάσαμε. Τώρα, η δική μου έκθεση τι επιδιώκει ε, θέλω να ακολουθήσουμε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να επαληθεύσουμε σε ποιο βαθμό οι καινοτομίε της συνθήκης της Λισαβόνας ε, έχουν ληφθεί υπόψη, υλοποιήθηκαν και σε ποιο βαθμό δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, ε, πρέπει να υλοποιηθούν ή πρέπει να τροποποιηθούν ενδεχομένως. Αλλά η φιλοδοξία μας πάει πέρα από αυτού. Πιστεύω ότι οι, οι διάφοροι κανόνες που αφορούν τα εθνικά κοινοβούλια στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπήκαν διαδοχικά, χωρίς να υπάρχει ένας πραγματικός σχεδιασμός, μια άποψη. Βεβαίως στο άρθρο 12 της Συνήκης Λισαβόνας αναφέρονται τα, τα καθήκοντα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχει αυτό το άρθρο, σύμφωνη, Αλλά δεν υπάρχει έτσι μια τακτοποίηση, ένα συστηματικό τρόπο παρουσίαση των καθηκόντων, αν θέλετε, των Εθνικών Κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να φτάσουμε σε μία ε, σύνοψη ε, για να ξέρουν πού να απευθυνθούν. Δηλαδή, σε τι αναφέρονται. Να έχουν και ένα σημείο αναφορά σε ένα μπούσουλα, αν θέλετε, τα εθνικά κοινοβούλια. Προφανώς είμαστε τώρα, έχουμε φτάσει σε κάποια φάση που είναι προσωρινή όμως. Πρέπει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε μια σαφή θεώρηση του στόχου μας ε, σε ό,τι αφορά την πλαισίωση των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ε, όλη διαδικασία. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένα γενικό προβληματισμό, ούτω ώστε να δούμε ποιος είναι ο τελικός ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και πώς θα ενσωματωθούν στο κοινοβουλευτικό ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει. Επίσης, το, τη σημασία των Εθνικών Κοινοβουλίων, τη μεγάλη σημασία, δεν την αναφέρει μόνο το άρθρο 12 τη Συνδίκη Λισαβόνα, που μιλάει για την ενεργητική συμμετοχή του στην ε, ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Αλλά προκύπτει η σημασία του και από κάτι πολύ απλό. Όταν ξεκινήσαμε την κοινοβουλευτική θητεία, ε, θέλαμε να σκεφτούμε ε, για την απόφαση του Ιουνίου του 2009. Θα θυμάστε ότι στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται ότι τα κοινοβούλια είναι οι κύριοι των συνθήκων. Είναι εκ των ουκάνευ αυτό. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε τα κράτη φυσικά, ούτε βεβαίως και τα κοινοβούλια τους, που είναι μια δημοκρατική διάσταση η πιο ας πούμε απτή των κρατών. Δεύτερον, Πάντα μιλάμε για τη γυπνίαση τη Ευρώπη με του πολίτε, για το πλησιασμά τη. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση, αυτή η λέξη. Τι σημαίνει ότι οι πολίτε θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, να είναι ενημερωμένοι, θα πρέπει να παθιάζονται με την Ευρώπη και φυσικά τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να βοηθήσουν και να κάνουν αυτή την, το πλησίασμα πολύ καλύτερα από εμά. Ε, Μερικέ φορέ γίνεται λόγο για την αντίστροφη επικουρικότητα. Δηλαδή, καταρχά, σε αυτό το επίπεδο την αρχική εξουσία, την αρχική αρμοδιότητα την έχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτή είναι η αντίστροφη επικουρικότητα. Δεν θέλω να σας απεικονίσω τώρα τη σημερινή κατάσταση. με τις καινοτομίες της συνθήκης της Λισαβόνας. Απλώς τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικοί εταίροι, σημαντικοί παίκτες. Επίσης θέλουμε να πούμε δύο λόγια για την πλαισίωση των Εθνικών Κοινοβουλίων, την ένταξή τους στο, στην κοινοβουλευτική ευρωπαϊκή διαδικασία. Κάποια από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι φυσιολογικές. Η συμμετοχή του Φερρυπίν, στην ε, διαμόρφωση των συνθήκων. Είναι προφανές αυτός. Άρθρο 48 Τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Συμμετέχουν και στη συνέλευση και συμμετέχουν στα πλαίσια της ε, επικύρωσης. Και στο άρθρο 49 που αφορά την ε, συμμετοχή και ένταξη νέων κρατών. Κάθε, με κάθε ας τροποποίηση των συνθήκων προφανώς εκεί εμπλέκονται και τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι προφανές. Αλλά κάτι που είναι πιο δύσκολο είναι να ενταχθούν τα εθνικά κοινοβούλια σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων τους. Μερικές φορές τα εθνικά κοινοβούλια έχουν την ε, δυνατότητα άμεσης ε, συνομιλίας με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Γράφεται στην συνθήκη ότι το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχουμε εμείς μόνο κατ' εξαίρεση, διάφορες ομάδες κρατών μπορούν να το ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος κανόνας βέβαια, αλλά Όταν εμείς είχαμε διαμαρτυρηθεί γιατί δεν είχαμε αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας, ε, είχαμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας αντίθετα το είχαν τα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχει μια άμεση σχέση, μια άμεση επαφή αν θέλετε. Ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια, την Κομισιόν και το Συμβούλιο, κάτι που εμείς δεν έχουμε. Δεν έχουμε αυτή την άμεση επαφή. Ε, και σε ό,τι αφορά επίσης την άσκηση του δικαιώματος ε, επικουρικότητας. Και εκεί υπάρχει άμεση αρμοδιότητα. Υπάρχουν άλλοι τομείς που τα Εθνικά Κοινοβούλια συνεργάζονται προφανώς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει το θέμα της ΚΟΖΑΚ, τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική. Τα όσα λέει το άρθρο 13 της Δημοσιονομικής Συνθήκης, συνεργασία πάλι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όλα αυτά τα περίπλοκα θέματα που μιλάνε για τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα έτσι διάχυτα. Το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται. Να φτιάξουμε ένα σωστό και αρμονικό πλαίσιο. Καταρχάς θα έχουμε ένα πιο ε, δημοκρατικό σύστημα. Με δύο σώματα. Με ε, μία εκπροσώπηση των ε, λαών και, μία, και ένα σώμα που, που εκπροσωπούνται τα κράτη. Παραδείγματο χάρη, ε, διάφορα ομοσπονδιακά κράτη, Ινδία, Βραζιλία, Ηνωμένε Πολιτείε, Ελβετία κτλ. Ε, έχουν το ομοσπονδιακό σύστημα, αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Όταν όμως εκπροσωπούνται με μοναδιαίο τρόπο ε, οι λαοί, Ε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες. Εμείς έχουμε το Συμβούλιο, ας πούμε. Εκεί εκπροσωπούνται τα κράτη, οι λαοί. Ε, το Συμβούλιο θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του δεύτερου σώματος. Σήμερα υπάρχει βέβαια η συζήτηση των κρατών στο επίπεδο του Συμβουλίου, αλλά μπορούμε όλα αυτά να τα συστηματοποιήσουμε περισσότερο. Τα κράτη εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Το θέμα της εκπροσώπησης των κρατών, ε, το σώμα το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη, μπορούμε όλα αυτά, αυτό το θέμα να το σκεφτούμε, να προβληματιστούμε από αυτού περισσότερο. Τώρα, Πώς θα δώσουμε προστιθέμενη αξία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα εθνικά κράτη ε, παίρνουν κάποιες αποφάσεις, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάποια πράγματα. Τι νόημα έχουν η Κομισιόν, το Συμβούλιο, η Κοζά κτλ αν δεν μπορούν να δώσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στοιχεία για να κάνει σωστά τη δουλειά του, να νομοθετήσει σωστά. Και από την άλλη, πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια όλα τα στοιχεία, ώστε να γνωρίσουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθε καλύτερα. Υπάρχει αυτή η δεύτερη διάσταση συνεργασίας σε συμβουλευτικό επίπεδο, ούτως ώστε να λειτουργήσουν με συμβουλευτικό τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια. Εντάξει, μερικές φορές γίνεται αυτό ad hoc, αλλά να γίνεται πιο συστηματικά θα θέλαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συνεχής πληροφορία, ροή της πληροφορίας, όπως ζητάει το άρθρο 12 της συνθήκης ούτως ώστε, προς τα κοινοβούλια, ούτως ώστε τα κοινοβούλια να παίζουν τον ενημερωτικό και πολιτικό τους ρόλο. Σε ό,τι αφορά αυτή την άμεση συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετέχουν ε, μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο στο Eurojust και στο Europol. Υπάρχει μια άμεση σχέση των Εθνικών Κοινοβουλίων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε επίπεδο Συμβουλίου και Κομισιόν και υπάρχει και μια οριζόντια σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μία επαφή προφανώς των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων με τους λαούς. και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να δείχνουν αυτή την ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δραστηριότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, για να διατηρούμε την επαφή με τους εκλογείς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σκεφτούμε τον θέμα του ελέγχου της επικουρικότητας και το θέμα της ΚΟΖΑΚ. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της επικουρικότητας, έχω την αίσθηση προσωπικά ότι χθε στην έκθεση του Γερμανού καθηγητή Μπερνής υπήρξε ένας σαφής ε, ορισμός της έννοιας της επικουρικότητας σε ό,τι αφορά την ε, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη συνεργασία δηλαδή της Εθνικής, των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν παίζουν το ρόλο της τροχοπέδης, αλλά συνεργάζονται ε, με θετικό τρόπο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διάφορες απόψεις που φτάνουν Ακόμη και αν δεν γίνονται κίτρινες κάρτες, ε, κόκκινες κάρτες, ακόμη και αν δεν μπλοκάρουν την ε, κοινοβουλευτική διαδικασία, αν τις λαμβάνουμε υπόψη, όπως πρέπει, η Κομισιόν, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, χωρίς κατά ανάγκη να προβούμε σε αυτό που ζητάνε, ε, υλοποιούν την άμεση συνεργασία. Οι γνώμες που φτάνουν, οι αιτιολογημένες γνώμες από τους πολίτες κτλ. Σε ό,τι αφορά τώρα τους, την Κοζάκ. Υπάρχει μια αμφισημία που πρέπει να ξεκαθαριστεί σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΚΟΖΑΚ. Είναι μια γενική λειτουργία αυτή ή ειδική αυτή της ΚΟΖΑΚ. Η ΚΟΖΑΚ προβλέπεται από τις συνθήκες, όπως ξέρετε. Είναι η μοναδική συνέλευση που έχει προβλεφθεί με οριστικό τρόπο. Γίνονται ψηφοφορίες προβλέπεται ο τρόπος ψηφοφορίας. Είναι ένα πράγμα διαρθρωμένο. Υπάρχουν όμως και άλλες διασκέψεις και άλλες ε, συνελεύσεις που εξετάζουν θέματα ασφάλειας, άμυνας ή οικονομικά θέματα. Επομένως, το θέμα είναι η ΚΟΖΑΚ, πιο συγκεκριμένα. Τι εξυπηρετεί. Στην έκθεσή μου θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Πρέπει να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε το σύστημα. Το προσπάθησα στην ομάδα εργασίας ε, που ασχολείται με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, βάζοντας όριο στις διακοινοβουλευτικές συνελεύσεις όχι πάνω από τέσσερις το μήνα. Να ξέρουμε σε τι, τι εξυπηρετούν, και επίση να αποφεύγουμε τι γενικόλογε συζητήσει, αλλά να επιδιώκουμε την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Η κόζα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να βλέπει πού έχει φτάσει, ποιο σημείο έχει φτάσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δηλαδή να, γίνει, να κάνει και μια γενική συζήτηση, αλλά και, και συγκεκριμένη, δηλαδή κάθε χρόνο κάνουν δύο, γίνονται δύο συνεδριάσεις, δηλαδή μία το εξάμεινο, και σε κάθε συνεδρία να, να λέμε να τα βήματα που έγιναν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ποια είναι τα εμπόδια, πώς τα ξεπεράσουμε, ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Γιατί αν δεν κάνουμε, δεν λειτουργήσει η Κοζάκ με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι χάνει την ιδιαιτερότητά της. Ε, εξομοιώνεται με άλλες μορφές διακοινοβουλευτισμού. Εγώ ανέφερα κάποιους προβληματισμούς. Φυσικά η, έκθεσή μου να προβαίνει σε πιο συγκεκριμένες σκέψεις, ιδέες και βεβαίως μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε θα ξεκαθαρίσω και τις δικές μου ιδέες. Και στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ που θα γίνει στην Αθήνα θα θέσω αυτά τα ερωτήματα. Και στα μέλη και στους προέδρους των διαφόρων εξειδικευμένων επιτροπών που ασχολούνται με ευρωπαϊκά θέματα και θα είναι παρόντες. Ε, θα του ζητήσω να μου πούνε τι ζητούν το καινούριο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Αυτά από μέρους μου και τώρα σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, thank you for... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. συζητούμε σύνθετα θέματα εκπροσώπησης, νομιμοποίησης, αποτελεσματικότητας, απόδοσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μέρος της πολυπλοκότητας αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα. Τα κοινοβούλια είναι πρωταγωνιστές και εμπλεκόμενοι στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε αλλά και στο εθνικό γίγνεσθε. Το ερώτημα κατά είναι πόσο έχει αποδώσει το σημερινό σχήμα. Υπάρχουν αιστείες τριβής. Αναφερθήκατε στην Κόζακ. Αρκεί όμως η Κόζακ. Αποδίδει. Εκπληρώνει τον ρόλο που υποτιθυρή είχε να λάβει. Η συνδίκη της Λισαβόνας βεβαίως ε, μας έχει δώσει ιδρυμένες αρμοδιότητες. Πράγμα όμως που ορισμένα εθνικά κοινοβούλια το θεωρούν ως ε, απώλεια δικών τους αρμοδιότητων και εξουσιών. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερο συντονισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συναφώς θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να μπούμε και στη θέση των εθνικών κοινοβουλίων για να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε τα της ενδεχομένης αντιπαλότητας μεταξύ των δύο. Πώς κατανέμονται, πώς θα έπρεπε να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου και αν υπάρχουν θέματα νομιμοποίηση επαναλαμβάνω και στα δύο επίπεδα. Κάτι το οποίο μας επαναφέρει στην ε, χθεσινή συζήτηση. Ως βάση θα μπορούσαμε να κινηθούμε με βάση την υπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση υλοποιείται σε δύο επίπεδα. Με όμω όμως, σε αρτήση του επίπεδου. Το τελευταίο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι το εξή. Χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση μεταξύ του εθνικού επίπεδου διακυβέρνηση και του ευρωπαϊκού. Μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων υπάρχει συγκυριαρχία, εκεί θα υπάρχουν τριβές και όσο θα υπάρχουν εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τα δύο αυτά επίπεδα να συνεργάζονται με τρόπο επικοδομητικό. Ευχαριστώ κύριο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σχήμα που μας παρουσιάσατε είναι πολύ ευρύ. Και εξάλλου το θέμα έχει πολλές πτυχές, πολλές πλευρές. Συμμερίζομαι και συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε. Συμφωνώ με πολλές από τις αξιολογήσεις σας και τις ιδέες σας. Να τονίσω ότι Έχει σημασία η χρονική στιγμή που υλοποιείται αυτή η έκθεση. Έχουμε λίγο χρόνο για να ολοκληρώσουμε αυτή την έκθεση. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να οριοθετήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα το αντικείμενο της έκθεσης, το θέμα της έκθεσης και να πιεστούμε, κατά την άποψή μου, να ξεκαθαρίσουμε, να διαφοροποιήσουμε δύο επίπεδα. Το επίπεδο το, της θεσμικής πραγματικότητας και των ρεαλιστικών τρόπων με τον οποίο εφαρμόζεται ή εφαρμόστηκε, εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται. Και ένα άλλο επίπεδο είναι το επίπεδο των αντιλήψεων που έχουν οι μεν και οι δε. σε πλαίσια μιας ιδεολογικής συζήτησης, στα πλαίσια μιας ανταλλαγής ιδεών που οδήγησε και σε, στις διάφορες συνθήκες. Μια συζήτηση που οδήγησε σε διαδοχικές συνθήκες, τροποποίηση συνθήκων κτλ. Είναι ένα πιο ευρύ θέμα, στο οποίο αναφέρθηκε ο προηγούμενος συνάδελφος και έχει και μια πολιτική διάσταση προφανώς. Και διαρωτώ πως αυτό το δεύτερο έχει νόημα το... να μην το εντάξουμε στην έκθεση και να ασχοληθούμε με τα όσα επιτάσσουν οι συνθήκες. Τα συνήθη θέματα, τα οποία παρότι δεν εξασφαλίζουν μια απόλυτη αρμονία, μια απόλυτη συμμετρία, Τελικά οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στα εθνικά κοινοβούλια είναι σαφείς, οριοθετημένες, με μία ή δύο μικρές εξαιρέσεις. Ο καθένας τελικά παίζει το ρόλο του. Για να υπάρξει δημοκρατική νομιμοποίηση των δράσεων των κυβερνήσεων. Ε, η μία από τις δύο, ένας από τους δύο τρόπους ε, νομιμοποίησης των ε, δράσεων είναι μέσω των κρατών. Με ένα πρόβλημα που αφορά το θέμα του του χώρου των ελευθεριών. Ακόμα και αν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις εξαιρέσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα τελικά. Ο καθένας ξέρει τις αρμοδιότητές του με βάση τα όσα επιτάσσουν οι συνθήκες. Γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στην εκπροσώπηση των πολιτών σε επίπεδο ένωσης, ποιος την εξασφαλίζει το Κοινοβούλιο, ε, που κάνει τον έλεγχο του προπολογισμού, τον δημοκρατικό έλεγχο και από την άλλη έχουμε τη λειτουργία, έχουμε την, την εκπροσώπηση των, κοινοβουλίων των ε, κρατών μάλλον, μέσω των εθνικών τους κοινοβουλίων. Παρότι δεν υπάρχει μια απόλυτη ενάργεια στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και ο κατάλογος του άρθρου της συνθήκης πραγματικά δεν εξασφαλίζει την απόλυτη ευκρίνεια, δεν είναι πολύ καρτεσιανός θα έλεγα. Παρόλα αυτά, Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο πώς λειτουργούν τα Εθνικά Κοινοβούλια σε αντιδιαστολή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά μιλάμε για το τρίτο σώμα, για, μιλάμε για την Αυτό το, αυτό το τρίτο σώμα θα είναι ένα σώμα συζήτησης. Τίποτε άλλο. Ένα φόρουμ συζήτηση. Και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια βέβαια είναι ο σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό τα μειώνει. Τα Εθνικά Κοινοβούλια από τη μία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άλλη παίζουν το ρόλο τους και συνεργάζονται, εξασφαλίζουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση, ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, μία ένας από τα φόρουμ αυτής της ανταλλαγής πρακτικών είναι η ΚΟΖΑΚ. Αλλά σε ό,τι αφορά το θεσμικό τους ρόλο, τον πολιτικό έλεγχο που ασκούν, τον έλεγχο των αποφάσεων κτλ. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα στις συνθήκες. Ακούσαμε κάποιες αφηρημένες ιδέες, εφάνταστες, ότι από αυτά τα νέα όργανα, από αυτές τις νέες έδρες ε, δημοκρατικής νομιμοποίησης, μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό ε, ε, είναι μια φαντασιοπληξία. Δημιουργούνται νέοι, νέα φόρουμ, ας πούμε, συνεργασίες, πράγματος χάρη για την ΚΠΑ, για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Μια άλλη διακοινοβουλευτική μορφή συνεργασίας προβλέπεται από το άρθρο 13. Όλα αυτά είναι διάφορα φόρουμ ενδιαφέροντα διαλόγου, χρήσιμα, που πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά δεν είναι εναλλακτική πόλη εκπροσώπησης της άσκησης της ε, κοινοβουλευτικής, ε, του κοινοβουλευτικού ελέγχου, διαφορετικής από αυτή που ασκούν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσοχή με όλα αυτά, έτσι. Και αμοιβαίο σεβασμό πρέπει να υπάρχει. Προσοχή και αμοιβαίο σεβασμό. Για να δούμε πώ θα προβούμε σε περαιτέρω βελτίωση, πώ θα βελτιστοποιήσουμε αυτές τις διακοινοβουλευτικέ μορφές συνεργασία χωρίς, κατά την άποψή μου, να υπάρχουν, να συντρέχουν οι λόγοι για να μπορέσουμε να διαβλέψουμε μια τρομακτική μεταρρύθμιση των σχέσεων Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτές οι ιδέες είναι ακόμα έτσι πολύ αδιαμόρφωτες, πολύ αφηρημένες ε, σε πολύ πρωταρχικό στάδιο. Ο κύριος Νταφ ζητάει το λόγο. Πρόεδρε, εν γέννη Συμφωνώ με την προσπάθεια επιτεύξης καλύτερης ποιότητας. Όμως, είναι πολύ νωρίες να αναθεωρήσουμε, να επαναξιολογήσουμε, αν θέλετε, τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις συνταγές της πίν όσον αφορά την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Γεγενεστέ. Είμαστε ακόμη στο πρώτο στάδιο. Ακόμη το πράγμα δεν έχει καθιζάνει, αν θέλετε, μετά την συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για στάδιο που χαρακτηρίστηκε από αποσπασματική λειτουργία και επηρεάστηκε τα μέγιστα από την ε, χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση. Θεωρώ συναφώς ότι θα αποτελούσε περιβολική διακινδύνευση το να ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Τον Μάιο έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Ξέρουμε ότι θα επικρατήσει πόλωση άνευ προηγουμένου μεταξύ φεδεραλιστών και οπαδών της επανεθνικοποίησης. Γνωρίζουμε επίσης τις ευαισθησίες ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά την εθνική κυριαρχία, ένα εξαιρετικά λεπτό θέμα. Ο κύριος Φόξ φιλοξενούνται πλέον αλλού, αλλά 95 συντηρητικά μέλη του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο ζήτησαν τα εθνικά κοινοβούλια να αποκτήσουν δικαίωμα αρνησικυρίας επί κάθε ευρωπαϊκής, επί κάθε ευρωπαϊκού νομοθετήματος. διάφορα πολιτικά κόμματα θα κατεβούν στον προεκλογικό αγώνα ζητώντα την ίδρυση ενός τρίτου κοινοβουλευτικού σώματος με τη συμμετοχή εθνικών βουλευτών σώμα το οποίο θα ελέγχει το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια, ένα δεύτερο σώμα, ένα δεύτερο κοινοβουλευτικό σώμα θα ελέγχει την λειτουργία του Συμβουλίου. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σκεφτούμε δύο φορές πριν ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Να σκεφτούμε λοιπόν οργανωμένα, προσεκτικά και να καταγράψουμε και τη θέση των εθνικών κοινοβουλίων επί του θέματος. Πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμπεράσματα ή τελικές αποφάσεις. Εξεπλάγει από αυτό που άκουσα ότι η συνεργασία, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν από το το της συνθήκης. και ότι πρέπει μετά το 2014 να παρέλθουμε ε, στο πλαίσιο μιας ε, διάσκεψης για να αναθεωρήσουμε τα πάντα. Όχι. Αυτά που είναι θετικά στην εκθέσή σα και πρέπει να ενθαρρύνουμε είναι τα εξή. Πρώτον, να ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο Υπουργών να δράσει σε περισσότερο θα λέγα κοινοβουλευτικό στυλ, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη διαβούλευση, περισσότερη συζήτηση. με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτικών απόψεων και των πολιτικών κομμάτων στις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Δεύτερον, όσο αφορά την ΚΟΖΑΚ, ετέθη το θέμα του κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πλήρη παρουσία στην ΚΟΖΑΚ. Ναι, πρέπει να είμαστε εκεί, πρέπει να είμαστε παρόντες, να μιλάμε, να συνεργαζόμαστε, Θα έλεγα, μάλιστα, επιπλέον, ότι είναι παράδοξο να συμμετέχει η αντιπροσωπεία μας στην ΚΟΖΑΚ στις αποφάσεις και μετά μας στέλνει σε εμά και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο ψηφίσματα Δεν νομίζω ότι συνάδει αυτό με το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άσε που δεν είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό. Να λοιπόν θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω στο πλαίσιο της συζήτησης για την εκθέσή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πιστεύω πως εργαστήκατε πάρα πολύ για να διαμορφώσετε αυτές τις ιδέες, να τις αποτυπώσετε και να διατυπώσετε τις προτάσεις σας. Χαίρομαι πολύ που άκουσα και τα δικά σας σχόλια και τα σχόλια των άλλων συναδέλφων τώρα όσον αφορά την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και την συνθήκη της Λισαβόνας. Δεδομένων των εξελίξεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για παράδειγμα, υπάρχει η επιθυμία να ενισχυθούν οι διακοινοβουλευτικές ε, σχέσεις. Αυτό φυσικά ε, είναι κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, συνάντηση το Δεκέμβριο με τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες και πιστεύω πως το ζήτημα είναι πολύ περίπλοκο και χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας στην έκθεση. Θεωρώ πως πρέπει να λάβουμε υπόψη από τη μία το πνεύμα της συνθήκης και τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά από την άλλη και τις αντιδράσεις για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα όσον αφορά την πρακτική συνεργασία. Επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι οι σχέσεις εθνικ... Ευρωπαϊκών κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αλλάξει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε υπολογίσιμη δύναμη και ορισμένα εθνικά κοινοβούλια δεν ε, είναι ευχαριστημένα από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζω την ιδέα του κυρίου Ντάφ για την Κόσακ, διότι πιστεύω πως πρέπει να κρατήσουμε τη παρούσα στάση και μια και είστε αντιπρόεδρος της Κόσακ, συμπρόεδρος μάλλον, πιστεύω πως έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία για το πώς θα γίνει αυτό και πώς η συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες ήταν εξαιρετική. Και είναι πολύ σημαντικό να ε, ετοιμάσουμε ένα, μια έκθεση με ένα σαφές και ξεκαθαρό μήνυμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την έκθεσή σας. Ο κύριος Χέφνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για την περιεκτικότατη εισαγωγή σας. Μας δώσατε τροφή για σκέψη σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μια που βρισκόμαστε στην αρχή λοιπόν, να αναφερθώ σε ορισμένα βασικά για μένα σημεία. Φαίνεται ότι είναι λογικό αυτή η έκθεση να εστιάσει έντονα στην στις παρούσες συνθήκες, στην παρούσα κατάσταση της συνθήκης της Λισαβόνας. Και να πω και εκ μέρους της κοινοβουλευτικής μου ομάδας ότι παρά τις δυσκολίες και παρά την αυξανόμενη απομάκρυνση από τον κοινοβουλευτισμό, σε πολύ σημαντικούς τομείς πολιτικής, η λύση δεν μπορεί να βρίσκεται σε πρόσθετα σώματα, σε επιπλέον βουλές οι οποίες θα συσταθούν και θα λειτουργούν μαζί με αυτό εδώ το κοινοβούλιο, με τα εθνικά κοινοβούλια που είναι άμεσα εκλεγμένα Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε αρκετά μακριά και αυτό φαίνεται και από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και από την δουλειά της Κόζακ και φυσικά υπάρχουν δυσαρέσκειες, σχετικά με το έργο της και πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Όμως πιστεύω πως μια αλλαγή των συνθήκων θα αποδυναμώσει το σύνολο των εργασιών μας, θα αποδυναμώσει αυτό το κοινοβούλιο και πιστεύω πως δεν είναι η σωστή λύση η δημιουργία επιπλέον σώματων και οργάνων. Είναι επίσης, ε, πιστεύω, ιδιαίτερα σημαντικά τα εθνικά κοινοβούλια, ο κοινοβουλευτικό έλεγχος που ασκούν στι κυβερνήσει τους, στο Συμβούλιο κατά επέκταση και το έργο το δικό μας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η δική μας ιδιότητα και εξουσίες ελέγχου που έχουμε. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η πρόταση θα αποδυναμώσει το έργο μας. Σημαντικό όμως είναι να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ουσιαστική συνεργασία Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την διαδικασία. Εγώ προσωπικά έχω συμμετάσχει στην ΚΟΖΑΚ, έχω συμμετάσχει πολλές φορές στις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και μετά από συνομιλίες και με ευρωβουλευτές και με βουλευτές, έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι η ικανοποίηση με την μέχρι τώρα συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων, παρότι υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν όμως πολλοί τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε, να προσανατολιστούμε καλύτερα. Πολύ συχνά ακούμε για τον έλεγχο για, την, τον έλεγχο που ασκείται μέσω της ε, ανταλλαγής απόψεων και θεωρώ πραγματικά περίεργο όταν κατά τη διάρκεια αυτών των δύο-τριών ημερών της κοινοβουλευτικής εβδομάδας καλούμε όλους αυτούς τους ε, βουλευτές, τους εθνικούς ε, βουλευτές, τους φέρνουμε στις Βρυξέλλες και τους καλούμε να μιλήσουν για την Τραπεζική Ένωση, για την Ευρωζώνη και από την άλλη εμείς έχουμε τις δικές μας ξεχωριστές συνεδριάσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν, συνεδριάσεις ε, οι οποίες είναι μόνο για εμάς και δεν έχουμε καμία επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως μπορούμε πρώτα να βελτιώσουμε την δική μας λειτουργία, το δικό μας τρόπο λειτουργίας. Τέλος, πιστεύω πως είναι λογικό, είναι συνετό και το άκουσα και από την ε, δική σας εισήγηση κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσει η εξέλιξη, η θεσμική εξέλιξη και στο τέλος να καταστεί δυνατός ένας ε, καλύτερος προσανατολισμός, μια καλύτερη οργάνωση όπως είπατε και εσείς, ένα δεύτερο σώμα, ένας καλύτερος ορισμός της νομιμοποιημένης συνεργασίας των θεσμικών οργάνων, των κοινοβουλίων μεταξύ τους. Όμως πρέπει πραγματικά να ξεχωρίσουμε τα πράγματα από την συνταγματική τους διάσταση και την ουσιαστική τους διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόνς είναι τώρα ο επόμενος φοιτητής. Ευχαριστώ. Αυτά που μας είπατε στην αρχή είναι αρκετά καθησυχαστικά, εκ πρώτης όψεως. Όταν αναφέρατε κυρίως τα σοφά τις ε, λόγια της ε, συνθήκης Λισαβόνας για τις αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν το λέω σαρκαστικά. Νομίζω ότι τα λέγατε πραγματικά ειλικρινά αυτά που είπατε. Αν είναι σαφέ ότι ο αριθμό των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αποκλειστικέ είτε επιμερισμένε, αυξάνονται και περισσότερο. Και μάλιστα μονοσήμαντα. τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα κράτη-μέλη ε, έχουν όλο και λιγότερες αποκλειστικές αρμοδιότητες. Δεν ξέρω αν την νομοθεσία μπορούμε να την προσμετρήσουμε και να την ποσοτικοποιήσουμε εύκολα ε, με μονάδες. Όλες αυτές οι νομοθεσίες που περνάνε τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μπορούν να συγκριθούν. Και η αναλογία των νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνάει η Ευρωπαϊκή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυξάνει εις βάρος των εθνικών νομοθεσιών. Και η πείνα που έχει η Ευρώπη για νομοθεσία δεν ε, κοραίνεται ποτέ. Οι αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων και των κρατών, επομένως, δεν μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στη σφετεριστή Ευρώπη δεν μπορούν να μεταφερθούν ξανά σε, εθνικό επίπεδο. Επομένω, τελικά, πού, τι γίνονται τα εθνικά κοινοβούλια. Γίνονται ε, συμβουλευτικά εκλεγμένα σώματα. Ε, σώματα όπως η ΚΟΖΑΚ είναι χρήσιμο. Είναι ένα από τα λίγα ε, θεσμικά όργανα που είναι χρήσιμα στην Ευρώπη. Αλλά δεν έχει εξουσία πραγματική. Συμβουλευτικό ρόλο έχει. Κάποια εργαλεία του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων όπως η επικουρικότητα, η αναλογικότητα κτλ. και το να εξετάζει ο σωστός φορέας ε, αυτό που πρέπει να εξετάσει με βάση τις αρμοδιότητες του, αυτές δεν είναι πραγματικές αρμοδιότητες. Η συνθήκη της Λισαβόνας για πρώτη φορά λέει ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να αποσυρθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό για πρώτη φορά λέγεται ρητά ε, και πάντα θεωρούσαμε ότι υπήρχε, μόνο που δεν το απεικονίζαμε σε καμία συνθήκη. Οι Βρετανοί συντηρητικοί είπαν ότι θα διαπραγματευτούν για να ξαναπάρουν κάποιες σημαντικές αξουσίες πίσω, σημαντικές για το εκλογικό σώμα. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι ποτέ δεν πρόκειται να τελεσφορήσουν τέτοιε διαπραγματεύσει και δεν γίνεται χωρί αλλαγή των συνθήκων με ομοφωνία για να μεταφερθούν αυτές οι αρμοδιότητες ξανά στο εθνικό επίπεδο. Το τελευταίο θέμα δεν σχετίζεται άμεσα με αυτό, αλλά όπως ο κύριος Νταφ, θέλω και εγώ να το συζητήσω. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των ε, ευρωπαϊκών εκλογών ε, σε ένα κλίμα πόλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σίγουρα θα έχουμε μία αυξημένη εκπροσώπηση του UKIP. Και αν νομίζετε ότι εγώ το επικυρώνω αυτό το κόμμα, ε, κάντε λάθος. Μάλιστα, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης δεν τους, κριτιμά, δεν τους κριτικάρουν. Καταρχάς, και στην Ολομέλεια ε, και στις επιτροπές ε, ελάχιστα βλέπουμε αυτούς τους κυρίους του, του UKIP. Και όμως αυτό δεν το λένε ούτε τα βρετανικά μέτρα, ούτε τα μέσα, ούτε τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Κάποιος είχε κατακεραυντώσει ας πούμε, τον κύριο Φάρας ότι δεν εμφανιζόταν ποτέ στις ε, συνεδριάσεις. Αλλά ποτέ δεν αναφέρθηκε ούτε στην Guardian, ούτε στον, στην Dependent, σε καμία εφημερίδα. το, η προβληματική συμμετοχή, για να μην πω το γεγονό ότι είναι εξαφανισμένοι αυτοί οι κύριοι. Σας ευχαριστώ για όλα, όχι μόνο για το τελευταίο που είπατε. Για τις παρατηρήσεις σας, για τις ερωτήσεις που κάνατε. Θα ακούσω και θα διαβάσω όλα αυτά που θα μου γράψετε. Θα ακούσω στην επόμενη συνεδρίαση και τους προέδρους της ΚΟΖΑΚ στην Αθήνα για να δω τι θα πούνε για αυτά τα θέματα. Όλες αυτές τις απόψεις θα τις εξετάσω. Κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι μπορείτε να πείτε τις απόψεις σας και έτσι να προσδιορίσουμε το θέμα, να το οριοθετήσουμε γιατί το θέμα είναι πολύ ευρύ. Μια αξιολόγηση που κάναμε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας που νομίζω ότι είναι και το αντικείμενο αυτή τη έκθεση είναι τι συμπληρωματικότητα πρέπει να πετύχουμε, τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να έχουμε ένα μπούσουλα για να το κάνουμε αυτό, για να το κάνουμε ποιοτικό τρόπο. Θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Σύστημα να πλαισιώσουμε, να εντάξουμε μάλλον και, το, και τα Εθνικά Κοινοβούλια, να δούμε τι ρόλο επακριβή παίζουν. Να γίνει μια συστηματοποίηση του ρόλου τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Ε, σε συνολικό επίπεδο, όχι σε κάθε τομέα, στο χ τομέα, στο ψ τομέα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να περιορίσουμε το θέμα και θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό, όπως είπε ο κύριος Χέφνερ. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν θέλουμε ένα τρίτο σώμα κοινοβουλευτικό. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα ανατρέπαμε και το σημερινό ε, σύστημα. Και επιπλέον ε, θα μιλούσαμε πολύ αφηρημένα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα. Γιατί για να υπάρξει τρίτο κάμερα θα πρέπει να υπάρχει και ένα δεύτερο σώμα που θα δίνει στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν το ρόλο της κυβέρνησης. Θα έχουμε δηλαδή τα, την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Εξάλλου, η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιγράψει με μηχανιστικό τρόπο τα σχήματα με τα οποία λειτουργούν τα εθνικά κράτη. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε καλά τα όσα λέει η συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να καταλάβουμε τι λένε τα κράτη. Αυτό που προκύπτει από όλα αυτά που ακούμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη συνεργασία των διαφόρων κρατών το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία, καλό είναι αυτό. Ωραία φράση. Αλλά τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Πώς θα είμαστε αποτελεσματικοί και πώς θα αυξηθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων χωρίς να αυξήσουμε χωρίς να ανατρέψουμε, χωρίς να αυξήσουμε, να μειώσουμε την αρμοδιότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μπρόνς, ας πούμε, δεν θέλει μεγαλύτερη εξουσία, περισσότερες αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, εγώ σας ευχαριστώ. Θα λάβω υπόψη τις ε, απόψεις και τους προβληματισμούς σας. Ελπίζω το συντομότερο να τον έχουμε ένα γραπτό κείμενο, ώστε να είναι και πιο συγκεκριμένη πρόταση και για να ακούσουμε μετά και τις δικές σας προτάσεις διόρθωσης, ε, βελτίωσης κτλ. Η, η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 10 Φεβρουαρίου, πολύ σύντομα λοιπόν. Και μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου σας προτείνω να παρουσιάσετε, σας προτείνω μάλλον ε, να περιμένετε τη γραπτή μου έκθεση η κυρία Γκουρμάη. Πιστεύω πως ε, είναι πολύ σημαντικό για όλους εσάς. Ναι, κάτι σύντομο. Είναι πολύ σημαντικό για όλους, πιστεύω. Ο κύριος Μαρτίνες έστειλε μια πρόσκληση για ένα συνέδριο σχετικά με την ε, εκδημοκράτηση. Και ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη θα είναι παρόν εκεί. Στις 2 Φεβρουαρίου, λοιπόν. Είναι, πιστεύω, σημαντικό. Μικρόφωνο. 22 Ιανουαρίου. Αύριο. Στη βιβλιοθήκη. Τι ώρα? Τι ώρα, λέει ο Πρόεδρος. 5.30. Πάμε τώρα στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που κανονικά έπρεπε να προηγηθεί της δική μου έκθεσης, το σημείο 9, που αφορά το ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικας. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή και το Δουνουτού. Σε ό,τι αφορά τις χώρες του προγράμματος της Ευρωζώνης. Ο κ. Σόλτς είναι ο εισηγητής. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε μία γνωμοδότηση που θα την υποβάλουμε στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Οικονομική Επιτροπή. Στι 11 Φεβρουαρίου θα υιοθετήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Παρακαλώ τον κύριο Σόλτ να πάρει το λόγο, να μας παρουσιάσει την εκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την κατανόηση και να σας ζητήσω συγγνώμη και για την αναβολή του θέματος αυτού, για την καθυστέρηση. Δυστυχώς ε, πρέπει να είμαστε πολλές επιτρόπες ταυτόχρονα και δεν γίνεται πάντα να είμαι στην ώρα του. Λοιπόν, η Οικονομική Επιτροπή έχει συντάξει μια έκθεση και εμείς έχουμε κληθεί να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με το ρόλο της ε, Τρόικας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η ε, Επιτροπή Απασχόλησης και Συνταγματικών Υποθέσεων, λοιπόν, θα συνοδεύσουν το έργο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή για να κάνουμε προεκλογικό αγώνα. Και οι δύο επιτροπές, αρμόδιες επιτροπές έχουν εισηγητές οι οποίοι ανοίγουν στις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν ορισμένες κριτικές, επικριτικές παρατηρήσεις στην έκθεση. Οι δραστηριότητες της Τρόικας έχουν γίνει αντικείμενο επικρίσεων από πολλούς διεθνείς οργανισμούς και από τους πολίτες, ιδιαίτερα εξαιτίας των μέτρων που έλαβε η Τρόικα στις ε, χώρες τις οποίες επενεύει. Ο Μάριο Ντράγκη το 2012, το, στο ζενίχ της κρίσης, είπε ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι παρελθόν. Και με αυτό εννοούσε την συνταγματική ασυμμετρία ανάμεσα στην οικονομική και την πολιτική διάσταση που επικρατούσε από τη συνθήκη του Μάστριχτ μέχρι τώρα. Στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης, το οποίο δυστυχώς δεν έπρεπε να ξεπεράσει τους 1500 χαρακτήρες, προσπάθησα να κρατήσω τις στο περιεχόμενό μου της αρμοδιότητας της Επιτροπής ΑΦΚΟ και να περιοριστώ στην σχέση ανάμεσα στα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στο Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήδη μόλις τώρα συζητήσαμε την πολύ περίπλοκη δομή των σχέσεων Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Πιστεύω πως καταρχάς χρειάζεται αποσαφήνιση στην ερώτηση του τι ακριβώς κάνει η Τρόικα και εάν έχει συνταγματικό δικαίωμα, αν υπάρχει νομική βάση για τη λειτουργία της. Η Τρόικα, όπως ζητήσαμε κι εμείς, πρέπει να είναι υπόλογη για το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θεωρώ πως δεν είναι. Φυσικά η Τρόικα έχει εξελιχθεί από τότε που δημιουργήθηκε. Ιδιαίτερα με την δημιουργία του μηχανισμού σταθερότητας. Έχει όμως εξελιχθεί σε ένα αυτόνομο όργανο το οποίο δεν βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και είναι μια μορφή συνεργασίας που βασίζεται σε μια εντολή που δεν προκύπτει από το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά από τον μηχανισμό σταθερότητας. στον οποίο συμμετέχουν και τα κράτη της Ευρωζώνης μέσω του Συμβουλίου του Μηχανισμού Σταθερότητας, του Συμβουλίου των Κυβερνητών. Κάτι το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάγεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν βασίζεται λοιπόν στο ευρωπαϊκό, στο κοινοτικό δίκαιο και συνεπώς δεν χαρακτηρίζεται από νομιμότητα. Σίγουρα θα θυμάστε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του συναδέλφου Μπροκ ότι απαιτήσαμε να δημιουργηθεί μια νομική βάση και εδώ παρατηρείται και η έλλειψη και οι λήψεις που υπάρχουν στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας και δεδομένων των εξελίξεων στα τέσσερα κράτη που στα οποία επενεύει η Τρόικα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία. Βλέπουμε ότι πρόκειται για χώρες της Ευρωζώνης. Μετά έχουμε τον μηχανισμό σταθερότητας, ο οποίος δημιουργήθηκε για τις χώρες της Ευρωζώνης ω ένα ε, μηχανισμό αντιμετώπιση και επίλυση ε, κρίσεων, ο οποίο όμως ε, δεν προκύπτει από το πρωτογενέ δίκαιο της Ένωση. Και είμαι πεπισμένο ότι η δική μας Επιτροπή θα έπρεπε να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα αναφερόμενη στην νομιμοποίηση και στην νομιμότητα του μηχανισμού σταθερότητας ο οποίος πρέπει να βασίζεται στο κοινοτικό δίκαιο και είναι ένα θέμα πολιτικής σημασίας. Θα χρειαστεί αλλαγή των συνθήκων και αυτό φυσικά πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια του, των συζητήσεων για το μέλλον της Τραπεζικής Ένωσης και της Νομισματικής Ένωσης. Στη γνωμοδότησή μου προσπάθησα να αναφερθώ και σε ένα επιπλέον σημείο της σχέσης ανάμεσα στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική σταθερότητα. Η κοινωνική σταθερότητα, ιδιαίτερα στις τέσσερις χώρες που αναφέρονται στην έκθεση, έχει άμεση σχέση με το έργο της Τρόικας. και οι προσπάθειες του Συμβουλίου να επιληθεί η κρίση εκτός κοινοτικού δικαίου δημιουργεί μια γκρίζα ζώνη νομοθετικά. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Επίσης, η γνωμοδότηση αναφέρεται στην αντίδραση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Κεντρικής Τράπεζας στην στα μέτρα. Ο συνάδελφος Σόπφλιν ήδη σήμερα το πρωί ανέφερε σε άλλο πλαίσιο βέβαια την ε, υπεροχή της πολιτικής έναντι στο δίκαιο και αυτό Θέλω να το επαναλάβω. Δημιουργείται, πιστεύω, το ερώτημα το του τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιδράσουμε πολιτικά έτσι ώστε να υπάρχει νομική βάση για τον μηχανισμό σταθερότητας. Αυτά που λέω δεν είναι από την σκοπιά της ε, πολιτικής μου ομάδας. Πιστεύω είναι χρόνος να ασχοληθούμε με το πρόβλημα αυτό, να επιληθεί το πρόβλημα αυτό της ε, νομιμοποίησης της Τρόικας. Διότι προκύπτει το ερώτημα και της ε, αντίδρασης των θεσμικών οργάνων. Εάν χρειάζεται κάποια αλλαγή των συνθήκων και το πόσο περίπλοκο είναι να γίνει αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει νομική βάση. Εγώ προσωπικά θεωρώ τη συνθήκη της Ελισαβόνας πολύ σημαντική και την ε, αντιμετωπίζω ως ε, σύνολο, ως ε, μια βάση και όσον αφορά το μέλλον και την ενίσχυση της ε, σύνθηκης αυτής που θα αποτελέσει τη βάση για, την, ε, για τις ε, μελλοντικές αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση κρίσης. Ο συνάδελφος Ελάινεν πρόσφατα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περισσότερη εξουσία από αυτή που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Μπαρόζο. Και σίγουρα οι αντιδράσεις της είναι πολιτικές, όμως έχουν και νομική διάσταση. Για εμένα δεν τίθεται μόνο θέμα διακυβέρνησης, αλλά είναι και καθήκον μας να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό πρέπει να γίνει μέσω του κοινοτικού δικαίου. Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος, διότι διαφορετικά παραβιάζουμε τα, τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά είπε ο συνάδελφος Λάινεν. αναφερόμενος και στις εξελίξεις που έγιναν στα τέσσερα, στις τέσσερις αυτές χώρες. Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου υπήρξε, υπήρξαν εξαιρέσει στην λειτουργία και στις εξουσίες που είχε η Τρόικα. Στην Επιτροπή μας ε, πιστεύω πως υπάρχει συμφωνία για το ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την κοινοβουλευτική εποπτεία. Αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πώς πρέπει να είναι δομημένος αυτός ο έλεγχος. Ευχαριστώ τους, διερμηνούς, τους διερμηνείς που μας, ε, θα μας δώσουν 10 ε, επιπλέον λεφτά. Έχω διάφορες που ζητάνε τον λόγο. Παρακαλώ σας ζητώ να κλείσετε το συντομότερο δυνατόν, ούτω ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε και στις ερωτήσεις που θα σας γίνουν. Σύντομα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μόλις θα ολοκλήρωνα. Είπα λοιπόν ότι θα υποβάλω τροπολογίες για να καταστήσω σαφές του ε, τι, προτείνω. Γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω εδώ και θα πω ότι θα χαρώ πολύ για την ε, καλή συνεργασία και τις τροπολογίες που θα έρθουν. Ε, να πρέπει να υπολογίσουμε το χρόνο. Σας παρακαλώ να μην μιλήσετε πάνω από δύο λεφτά. Αν φύγουν οι διερμηνείς, θέλω να σας πω πριν φύγουν οι διερμηνείς, ότι μέχρι τις 23 Ιανουαρίου το, στις 12 το βράδυ, πέμπτη, μέρα πέμπτη, μπορείτε να παρουσιάσετε τις τροπολογίες σας. Ο κύριος Σέφλιν. Πρόεδρε, μια συγκεκριμένη απάντηση προς τον κύριο Σούλτς. Η θέση μου έχει ως εξής. Χωρίς πολιτική συνένεση, ένα πολιτικό πλαίσιο είτε αποδίδει είτε έχει μόνο αρνητικές τα λειτουργεί αρνητικά μετά ένα από τα κύρια προβλήματά μας είναι ότι το έργο της Τρόικας είναι εξαιρετικά τεχνικό, εξελίσσεται κρυπτό και είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Συμφωνώ κρετάλα ότι επλήγησαν οι πολίτες λόγω της λειτουργίας της Τρόικας. Δεν υπήρξε διάλογος σε διάφορα επίδεξουσία και θα έλεγα επίσης ότι αν μπορεί φαίνεται όλα αυτά προέκυψαν υπό την πίεση των γεγονότων. Πρόκειται για μια παγκοσμία απειλή, αλλά αυτό αφορά μόνο το βραχυπρόθεσμο. Τελείωσε όμως το βραχυπρόθεσμο. Και αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέτε, αυτό τελείωσε. Αυτό λέτε κι εσείς. Πέραν αυτού όμως έχουμε το θέμα της λογοδοσία Ορθών. Δεν διαφωνεί κανεί. Το πώ θα αποκατασταθεί η λογοδοσία το τονίζετε κι εσεί στο αρχικό σα κείμενο. Και πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο πλήττει την δημοκρατία εν τέλει. Αν δεν ε, τεθούν όλα αυτά υπό επαρκή δημοκρατικό έλεγχο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράνγκελ έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς. Να αποδεχθούμε ότι αυτό ήταν μια κατεπίγουσα λύση, ότι δεν υπήρχαν όργανα, μηχανισμοί, ένα, ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Να το τονίσουμε αυτό λοιπόν καταρχά. Δεύτερον, να πούμε επίσης, ιδιαίτερα επειδή συζητούμε αυτές τις μέρες και το θέμα των Εθνικών Κοινοβουλίων, να πούμε λοιπόν έλεγα ότι στις τέσσερις χώρες με πρόγραμμα στήριξης με Τρόικα, με Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο έγιναν εθνικές εκλογές στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Άλλαξαν οι κυβερνήσεις. Όλα τα κόμματα συμμετέσχουν στις διαπραγματεύσεις. Το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα εν μέσω της διαδικασίας και έγινε και στην Κύπρο. Αλλαγή πρόεδρου είχαμε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει νομιμοποίηση, δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας σε εθνικό τουλάχιστον επίπεδο, σε εθνικό πλαίσιο. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Αυτά δεν έγιναν στην πλάτη των λαών. Έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη τους. Μπορεί να υποφέρουν. Μπορεί να είναι κατά πολλών μέτρων, εν τούτης, ψήφισαν υπέρ των συγκεκριμένων κομμάτων που υποστήριξαν το πρόγραμμα στήριξης και την εφαρμογή του. Δεν λέω ότι συμφωνώ με τα προγράμματα, άλλωστε συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις σας στην έκθεση. Όμως, ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι σημαντικές πλειοψηφίες τάχθηκαν υπέρ εν τέλει των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η σχέση κειμένου του κυρίου ε, Σόλτ θα πρέπει να εμπλουτιστεί και να ξεκαθαριστεί σε ένα τομέα κυρίως όπου υπάρχει και το βασικό έλλειμμα της, ε, του κειμένου της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα αυτό το νομικό θεσμικό παζλ που βρίσκεται πίσω από το σύστημα της Τρόικας και που μετά την έγκριση του δίπτυχου καονισμού του Τούπακ, το παζλ αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε την αρχική απόφαση για τη δημιουργία του EFSF, του Ευρωπαϊκού Ταμείου δηλαδή ε, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ε, συνεχεία το θέμα των ε, διμερών δανείων για την Ελλάδα. συνεχεία, το Μάιο δημιουργεί ένα διακυβερνητικό σύστημα κοινό ε, με δάνεια υπό προϋποθέσεις. Έχουμε το άρθρο της συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 13-16 μέσα σε ένα πιο διακυβερνητικό πλαίσιο και παράλληλα όμως έχουμε τη συνθήκη του ESM και μετά υπάρχει και το 2 με ένα σύστημα ενισχυμένης εποπτείας από την Κομισιόν για τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια. Αυτά τα τρία επίπεδα δεν είναι πια συμβατά μεταξύ τους. Πέρα από τις πιο ριζοσπαστικές λύσεις που αφορούν την μεταρρύθμιση των συνθήκων και του άρθρου 143, εγώ νομίζω ότι ήδη στα πλαίσια των σημερινών συνθήκων, λόγω των αντιφάσεων που υπάρχουν μέσα στα διάφορα διαφορετικά αυτά νομοθετικά επίπεδα και των αποφάσεων των κρατών μελών ή των διεθνών συνθήκων, πρέπει να ξεπεράσουμε το μηχανισμό της ε, Τρόικας. Είναι αναγκαίο αυτό. Ή να εντάξουμε τα, τις αρμοδιότητες της Τρόικας μέσα στο ενωσιακό πλαίσιο, στο νοσιακό θεσμικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Χέλμου τσόλτ για τη γραμμοδότησή του, η οποία είναι πολύ σύντομη και περιεκτική και έτσι έπρεπε να είναι και παρότι είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Πρέπει να πούμε ότι ήταν έκτακτα μέτρα. Δεν ήταν τίποτα άλλο. Όμως δεν μπορούμε να πάρουμε μια ενδιάμεση λύση, μια προσωρινή λύση και να τη μονιμοποιήσουμε. Σε τέτοια περίπτωση τότε θα οδηγηθούμε σε μια Ευρώπη η οποία δεν θα είναι εκλεγμένη, δεν θα είναι δεν θα έχει νομιμότητα, δεν θα έχει την ε, πολιτική ευθύνη που πρέπει να έχει, αλλά θα είναι μόνο ένα όργανο γεμάτο γραφειοκρατία. Και πρέπει πραγματικά να αναλογιστούμε τι σημαίνει όλο αυτό για τους πολίτες μας. Πιστεύω πως η έκθεση ε, πρέπει να δείχνει ξεκάθαρα την διάσταση αυτή, πρέπει να δείχνει την δυσαρέσκεια που υπάρχει για αυτό το ε, σύμφωνο, για αυτή την παρέμβαση της Τρόικας στην Ευρωζώνη. Τώρα όσον αφορά τα, ζητήματα, δημοσιονομικά ζητήματα, τα συνταγματικά ζητήματα και αυτά επίσης πρέπει να έχουν νομικότητα, πραγματικά, νομιμότητα. Πραγματικά αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη διάσταση θα φύγουμε πάρα πολύ, θα απομακρυνθούμε πάρα πολύ από το σκοπό μας. Και πραγματικά ανησυχώ για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως αυτό εξελίσσεται. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση, η γνωμοδότηση Σόλτς και ανυπομονώ να παρακολουθήσω και να συμμετέχω στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Γρήγορα να απαντήσει ο κύριος Σόλτς, παρακαλώ. Πιστεύω πως από τη συζήτηση φάνηκε ότι είναι μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση και είναι πολύ σημαντικό το να δούμε, το να απαντήσουμε στο αν μπορούμε πραγματικά να δικαιολογήσουμε τις ενέργειες κάποιου μέσου που έχει συσταθεί προσωρινά και για, έκτακτους, για έκτακτες περιπτώσεις. και να σας παραπέμψω στον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της ε, Γερμανίας. Σύμφωνα με τον οποίο ο πρόεδρος της Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, έχουν ξεκάθαρη εντολή. Η Τρόικα όμως όχι. Λείπει η βάση. Η βάση που προκύπτει μόνο από τις συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρέπει να προσπαθήσουμε στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων να δώσουμε την συνταγματική διάσταση και να αναφερθούμε ιδιαίτερα σε αυτό, σε αυτή την συνταγματική βάση, νομική βάση και να κερδίσουμε έτσι ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. 23 Ιανουαρίου μέχρι τις 12 το βράδυ για τις τροποποίησεις. Ο κύριος Τάραντ θα μπορούσε να μιλήσει παρακαλώ πολύ σύντομα. Ήθελε να κάνει μια δήλωση. Thank you, Mr. President. Πρόεδρε. Ένα μισή λεπτό. Κοιτάξτε, όταν κάποιος φεύγει, πρέπει να συνεχίζουμε την κληρονομιά που μας άφησε πίσω του Μιλώ για τον κύριο Τσαρκόφσκι για την, για την εκθεσή του. Δεν καταρθώσαμε να εξασφαλίσουμε επαρκή υποστήριξη, αρκετές ψήφου λόγω της απουσίας του στη Σιβηρία. Εν πάση περιπτώσει, να μην αφήνουμε πράγματα στη μέση. Να συνεχίσουμε με γραπτές δηλώσει. ή να πάρουμε μια απόφαση να τα ξεχάσουμε όλα. Πήραμε μια απόφαση πριν από λίγο καιρό. Και Γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι όταν μια γραπτή δήλωση κάποιου βάρου μένει στη μέση δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ διαβάζω ο κ. Μπροκ και 11 βουλευτέ ξεκίνησαν μια γραπτή δήλωση για του κινδύνου του εθνικισμού, του αντισημιτισμού και άλλων μορφών εθνική μυσαλλοδοξία. φτάσαμε ξαφνικά στις 150 ψήφους ε, και δεν λέω με αυτό ότι είναι αντισημιτικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως οι συντονιστές και άλλοι έχουν ευθύνη. Πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα και να κάνουμε μια, να κάνουμε μια πρόταση, να τελειώνουμε με αυτό, να μην αφήσουμε στη μέση ε, αυτή την γραπτή δήλωση, γιατί νομίζω ότι ε, είναι παράδεκτο το καταγράφουμε. Καταγράφουμε αυτό το σχόλιο σας. Πρέπει να κλείσουμε πια τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πρώτα ξανά του ε, διερμηνείς για τον επιπλέον χρόνο που διαθέσαμε. Γεια σας, ευχαριστώ.